με βάση τον νόμο και την τρομοκρατία ε, εκτεί την ποινή του. Φαντάζομαι θα θέλατε να μην είχε δικαστεί ποτέ. Αυτό θα θέλατε. Ευχαριστώ. Όχι, όχι. Έκλεισε η συζήτηση τώρα. Και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση κλούνα για την υιοθέτηση από την Εστονία του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2011. Ε, στρέφομαι καταρχάς προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Σεκλούνα, για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ευτυχής που μπορώ να παρουσιάσω αυτή την έκθεση και την αίτηση της Εστονίας να γίνει μέλος της Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται ένα κράτος και χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοια δύσκολη επαφή. Αυτό λέει πολλά για τη χώρα, για την Ευρωζώνη και για το ευρώ. Ο λόγος για τον οποίο ζητούμε να προσχωρήσουμε στο ευρώ είναι διότι η Εστονία έχει σεβαστεί τα κριτήρια του Μάστριχτ και τα επιτεύγματα αυτά επετέχθησαν στην χειρότερη χρηματοοικονομική κρίση και κοινωνική κρίση που έχουμε διαπιστώσει στη διάρκεια ζωής μας και ε, υπάρχει μία συνεχής και αξιόπιστη προσπάθεια της ιστορικής κυβέρνησης και του λαού και η κοινή γνώμη παρόλα τα προβλήματα είναι υπέρ του να προσχωρήσει στο ευρώ. Ε, σαν εισηγητής έχω έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση, με την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όταν δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση συγκλήσεως. Ε, συζήτησα με όλους και αντιλαμβάνομαι ότι τα επιτεύγματά μας είναι προς τιμήν της χώρας μου. Αλλά είχαμε ελάχιστο χρόνο για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσει την έκθεσή του μετά από την δημοσίευση της εκθέσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι είναι απερκής ο, ο, χρόνος και δεν ε, ε, σεβόμαστε το Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Ε, γι' αυτό και... Ε, δώσαμε μία προφορική εξήγηση ε, της πρόοδου μας. Ελπίζω όμως ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη αυτής της διαδικασίας όταν θα υπάρξει άλλη υποψήφια χώρα. Και κατά τη γνώμη μου, εάν ακολουθούσαμε αυτή την ε, λύση ε, δεν θα ήταν προς όφελο της Ευρωζώνης. Ε, θέλουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και εμείς το ευρώ στη δύσκολη αυτή εποχή διότι διαφορετικά κανείς δεν θα βοηθηθεί στη δύσκολη αυτή περίοδο. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα για να μπορέσει να υπάρξει βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μέτρων και κατά τη γνώμη μου η Εστονία θα αποτελέσει ένα προσόν για την Ευρωζώνη και ήδη το, στο τέλος του 2009 είχε το χαμηλότερο έλλειμμα του δημοσιονομικού προϋπολογισμού σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το γεγονός λοιπόν ότι καταφέραμε τις, τα καλά έτη να δημιουργήσουμε πλεονάσματα οδηγεί ε, σε πολλούς, πολύ καλούς δείκτες της ε, χώρας και παρόλη την ε, δύσκολη κρίση μπορέσαμε να κρατήσουμε σε καλή τάξη τα οικονομικά μας. Είμαστε μία από τις χώρες η οποία φορολογικά είναι πολύ πειθαρχημένη και γι' αυτό και έχουμε βιώσιμα ε, δημοσιονομικά στοιχεία και η αίτηση της Ιστονίας είναι ένα σύμβολο για τους γείτονές της ότι η προσχώρηση στο ευρώ θα είναι μία ευχάριστη λύση για αυτούς που έχουν προετοιμαστεί και τέλος δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μία εύκολη πορεία μπροστά για την Εστονία διότι η ανεργία είναι πολύ υψηλή και ο κίνδυνος πληθωρισμού δεν ε, είναι πουσιώδης και για το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής και υποβάλλω προς εξέταση στο Κοινοβούλιο αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Ρέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έντουαρτ Σκυκλούνα για την πολύ ισορροπημένη ουσιαστική έκθεσή του για την ε, σύγκληση και για τη, της και την ε, προσχώρησή της στη ζώνη του ευρώ. Είναι σημαντικές οι προσπάθειες που κατέβαλε η Εστονία για να φτάσει σε αυτό τον όρο σταθμό. Και πιστεύω ότι όλοι υποστηρίζουμε τις ε, προσπάθειες ε, της ε, Εστονία για ένταξη στο ευρώ. Και έτσι η πρόταση της Κομισιόν μετά την 20 Ιουνίου πρέπει να πάει ακόμη πιο πέρα και να καλωσορίσουμε την Εστονία στη ζώνη του ευρώ την προσεχή, την η απόφαση για την έγκριση του ευρώ από την Εστονία θα γίνει έχοντας ως υπόβαθρο πολύ χαλεπούς καιρούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως τους χαλεπέστερους από ιδρυσεώς της. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, η θετική αυτή αξιολόγηση για την Εσθονία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σήμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που εκπέμπουμε για να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρω λειτουργική. Τονίζεται επίσης ότι σε αυτή την εκτίμηση που γίνεται. Τα κράτη-μέλη εξετάζονται και αναλύονται με βάση τις επιδόσεις τους, με βάση τα πλεονεκτήματα, τα υπέρτα κατά και με ίσους όρου, με ισότιμη μεταχείριση. Η θετική λοιπόν αυτή η εκτίμηση για την Εστονία είναι και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που εκπέμπουμε προς τις αγορές αλλά και για την ε, ζώνη εκτός, ε, για τα κράτη-μέλη εκτός ζώνης ευρώ υπό την ε, παρούσα συγκυρία. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Εστονία θα προσχωρήσει στο ευρώ έχοντας βρισκόμενη σε ισχυρή θέση με πολύ αξιόπιες πολιτικές, έχει πολύ καλή φορολογική θέση, έχει πολύ χαμηλό επίπεδο ελλείμματος. While the average in the European Union is uh, currently το 75% συνήθως είναι το έλλειμμα, το δημόσιο έλλειμμα στην Ευρώπη, στη ζώνη του ευρώ. 7,2 μόνο είναι στην Εστονία. Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για τεράστια διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο. Σίγουρα δεν ε, είναι δεν θα βγει αλόβητα από αυτή την κρίση και η Ιστονία, αλλά αλλά από το 1992 και μετά και για δύο δεκαετίες έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Η έγκριση του ευρώ λοιπόν δεν νομίζουμε ότι θα οδηγήσει σε, σημαντική, σε σημαντικές αναταραχές και διαφορές. Βέβαια, η έγκριση του ευρώ δεν θα είναι και ο τελευταίος σταθμός. Το αντίθετο, αν εγκριθεί, στην, αν υιοθετηθεί το ευρώ του χρόνου στην Εστονία, θα πρέπει να παραμείνει η πειθαρχία στις πολιτικές και θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, πολιτικές στον τομέα το δημοσιονομικό, τον εποπτικό, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις στις χώρες εντός της ζώνης του ευρώ. Και ρετίζω την προθυμία των αρχών της Εστονίας να εξασφαλίσουν με επίσημη επιστολή που έστειλαν ε, στις χώρες μέλη του ευρώ ότι δεσμεύονται να τηρήσουν τις πολιτικές της ε, ζώνης του ευρώ και να θεσπίσουν και τις ανάλογες εθνικές πολιτικές. Παραλλήλως βέβαια είναι απαραίτητο η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη να ενισχυθεί. Οι πρόσφατες προτάσεις της Κομισιόν και για την εμβάθυνση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και για την διεύρυνση της ζώνης του ευρώ με βάση επιδόσεις των χωρών το καταδεικνύουν. Ο στόχος μας είναι μια ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική οικονομική και νομισματική ένωση. Κύριε Πρόεδρε, ξεότιμοι βουλευτές, για να ολοκληρώσω, μετά τις ε, διαβουλεύσεις που είχαμε αυτή την εβδομάδα, που θα έχουμε μάλλον αυτή την εβδομάδα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ακολουθήσει συζήτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αργότερα, αυτή την εβδομάδα. Και αν όλα πάνω όπως ε, υπολογίζουμε θα εγκριθούν όλες οι σχετικές νομικές πράξεις ε, μέχρι το Συμβούλιο της 13ης ε, Ιουλίου, κάτι το οποίο θα δώσει επαρκή χρόνο στην Ιστονία να προετοιμαστεί για τη μετάβαση και για την υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, πολλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις προτάσεις σας και να συγχαρώ θερμά Ευχαριστώ. Και τώρα οι πολιτικές ομάδες, ο κ. Μίτσελ από το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια έκθεση. Ε, την υποστηρίζω. Ε, υποστηρίζω τη γενική ιδέα και τα γενικά του σχόλια και τις ανησυχίες που μας ε, κοινοποίησε. Θα ήθελα να σας πω ότι Είμαστε σε θέση να δεχθούμε την Εστονία στο χώρο του ευρώ λόγω των θυσιών που έκανε ο εστονικός λαός και την ισχυρή ηγεσία του Κοινοβουλίου και της ε, κυβέρνησης. Αυτή η ηγεσία ξεπερνάει την απλή πειθαρχία των δημοσιονομικών και την ε, πρόθεση των ε, θυσιών. Ε, υπήρξαν μεγάλες αβεβαιότητες για το μέλλον ε, και ανησυχούσαν για την Ευρωζώνη διάφοροι. Ε, και εν μέσω ανησυχιών ε, αυτή η μικρή χώρα μας δείχνει το δρόμο. Είναι φάρος όχι μόνο για τις χώρες στην περιοχή αλλά για όλη την Ευρώπη προκειμένου να υπάρξει μια αναζωογόνηση της εμπιστοσύνης μας σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τους, στους βουλευτές ότι τα πρώτα δέκα χρόνια του ευρώ 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ περισσότερες ε, από ό,τι στις είπα την ίδια εποχή. Ε, μία ε, θαραλέα λοιπόν κυβέρνηση ε, και ένα θαραλέο κοινοβούλιο πέτυχε αυτό που πέτυχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που πέτυχε και θα είναι αποφελές για αυτή τη μικρή χώρα, όπως είναι και για τη δική μου, που είναι επίσης μικρή χώρα. Για να σκεφτούμε λοιπόν το εξή. Αυτέ οι μικρέ χώρε, πού θα είμαστε αν δεν είχαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν και τους, τους υπουργούς οικονομικών στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ σε αυτές τις δυσκολε στιγμές. Ε, θα ήθελα να μιλήσω για αυτόν τον κύκλο άνθησης και ύφεση που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και το, το θέμα του πολλαπλασιασμού των τίτλων και αξιογράφων για τον οποίο, θέμα για το οποίο δεν μιλήσαμε. Θα πρέπει να δούμε πώς τα χαμηλά επιτόκια και ο χαμηλός πληθωρισμός ε, μας ε, οδηγεί σε μια κατάσταση ε, πολλαπλασιασμού των τίτλων και αξιογράφων. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Είναι μακρά η νύχτα. Γι' αυτό θα είμαι αυστηρή μαζί σας. Ο κύριος Πάντα ε, από του Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Την Τετάρτη θα ψηφίσουμε για την ε, έκθεση ε, με σκοπό να ενταχθεί η Εστονία στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει να περιμένουμε περίπου ένα μήνα για την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου. Η υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία είναι ακόμη ένα βήμα στην διαδικασία ολοκλήρωση. Είναι φυσική διαδικασία μια συνετού δημοσιονομική πολιτική που έχει η Εσθονία επί χρόνια. Ήδη στις αρχικές στιγμές της οικονομικής κρίσης, εμείς καταλάβαμε ότι οι προκλήσει της κρίσης απαιτούσε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και ένα νέο προβληματισμό ε, και ανασχηματισμό παλιών πολιτικών. Μια νέα προσέγγιση οδήγησε σε πολλές δημοσιονομικέ. Ε, περικοπές το 2008 και 2009. Η υιοθέτηση του ευρώ σημαίνει ότι οι προσπάθειές μας δεν ήταν εισμάτη. Όλες οι εξελίξεις του περασμένου έτους δείχνουν τη σημασία των αξιόπιστων στατιστικών και την αποφυγή των δαπανών. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την ε, συνετή αυτή δημοσιονομική πολιτική είναι πολύ σημαντικό αυτό το ευρώ δηλαδή για μια μικρή και ανοιχτή οικονομία. Δεν υπάρχει ανεναλλακτική λύση. Επίση, ε, η υιοθέτηση του ευρώ από την Εστονία είναι θετικό βήμα και για την Ευρώπη. Η πίστη μα στην Ευρώπη μοιάζει με την έξοδο από ένα μακρύ μαύρο τούνελ. Νομίζω ότι όταν δεχτείτε την Εστονία ε, στην Ευρωζώνη θα δεχτείτε ένα μέλος το οποίο καταλαβαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα ενδυναμώσουμε την ε, ΟΝΕ και το ευρώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφου, τον εισηγητή τον κύριο Σκυκλούνα και τους κοιόδης εισηγητέ για την εποφελή συνεργασία. Σας διαβεβαιώ ότι είμαστε έτοιμοι για την προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Και τώρα ε, από την ομάδα των φιλελευθέρων ο κύριος Κλίντς για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, Όντως από το, ε, ε, την 1η Ιανουαρίου του χρόνου το 17ο μέρος της ε, Ευρωζώνης θα είναι η Εστονία και πρέπει να τους συγχαρούμε για το θάρρος τους διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι οι υπεύθυνοι έκριναν ε, σωστά και δεν ε, πρόθυσαν πολιτικές σκοπιμότητες και ε, αντιλαμβανόμαστε την τρομερή προσήλωση και θέληση και προσπάθειες της χώρας που κατάφεραν υπό αυτά τις προϋποθέσεις να καλύψουν τα αναγκαία κριτήρια και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν παραμείνει προσιλωμένοι ή στις επιταγές της συνθήκης και θέλουν ε, ε, να προσχωρήσουν γρήγορα. Αυτό με ικανοποιεί γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ακόμη χώρες οι οποίες ε, έχουν εμπιστοσύνη στην κατάσταση της κοινότητας και αντιλαμβανόμαστε ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανήσυχοι. Βλέπετε ότι το ευρώ έχει προβλήματα προβλήματα και στην χώρα φοβούνται ότι θα ακριβίνει η ζωή με την εισαγωγή του ευρώ όπως έγινε στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και ε, σαν μέλος της Ευρωζώνης θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει και τα θέματα των χρεών της Ευρωζώνης. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να μας διευκρινίσει ορισμένα σημεία. Ελπίζω ότι η μελλοντική ε, πορεία θα είναι θετική και θα μπορέσει να είναι και βιώσιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα η κυρία Σφίνμπερν για 1,5 ε, λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σικούνε για την σαφή έκθεσή του. Στηρίζουμε την προσπάθειά τους διότι σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών ταραχών χάρη στι τις δημοσιονομικές δεξιότητες της χώρας κατάφεραν να, να καλύψουν τις προποθέσεις προσχώρησαν και πρέπει να τους επιβραβεύσουμε διότι εάν ένα κράτος μπορεί να εφαρμόσει τα αυστηρά κριτήρια σε αυτές τις δύσκολες εποχές θα πρέπει ε, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους πολίτες της χώρας αυτής. Ο κύριος Μπρόντς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να συγχαρούμε την Εστονία. Εγώ θα τους λυπόμουν και θα τους έδινα τα συλληπιτήριά μου. Διότι πρέπει αυτό να έχει σχέση με την σχετική κίνηση εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων και με τις ανάγκες. Διότι αν δεν καλύπτει τις ανάγκες της οικονομίας της θα διαπιστώσει ότι όλα τα προβλήματα θα χειροτερεύσουν και αυτό διαπίστωσε και η Μεγάλη Βρετανία όταν ήταν μέλος του συστήματος συναλλαγμάτων και μπορέσαμε να ε, γλιτώσουμε μόνο όταν εγκαταλείψαμε ε, το σύστημα ε, του ευρωπαϊκού συναλλάγματος. Τώρα υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που ελοχεύουν και ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θέσουν πολύ ψηλά την ε, συναλλαγματική τιμή της ε, κορώνας με το ευρώ και ε, τότε θα υπάρξει μία πτώση του ισοζυγίου πληρωμών. Το, η Εστονία θα χάσει την κυριαρχία της ε, οικονομικά και άρα και πολιτικά και είναι ηρωνικό διότι είναι μια χώρα η οποία ξέφυγε από τα δόντια του κομμουνισμού μόνο πριν από 19 χρόνια. Οι επιμέρους ομιλητές τώρα. Εμείς όταν είμαστε φύλαχλοι περιμένουμε να έχουμε μια ομάδα που να έχει καλή πειθαρχία και όταν παίζει καλά και έχει πειθαρχία, κανονικά θα κερδίσει στο παγκόσμιο κύπελο. Ε, αυτό το κανόνα θα πρέπει να το εφαρμόσουμε και για τη διεύρυνση του ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα βραβείο για τη δημοσιονομική πειθαρχία και για τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες προβαίνει κανείς. Όταν υπάρχει ύφεση ε, μεταξύ του, δηλαδή, του 2005 και 2008, κατά την περίοδο της ύφεσης, τα περισσότερα κράτη-μέλη ξόδεψαν πολύ περισσότερο από το δυνατό και το πρέπον. Νομίζω όμως ότι οι Εστονοί φίλοι μας ήταν πιο έξυπνοι. Ε, αντί να δαπανίσουν, δημιούργησαν αποθεματικά στον προϋπολογισμό. Χάρη σε αυτά τα αποθέματα, χάρη στον προϋπολογισμό τους, η ύφεση το 2009 δεν οδήγησε σε καμία χειροκοπία στη χώρα. Με χάρη σε αυτή την ε, αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, η Εστονία κατάφερε να σεβαστεί όλα τα κριτήρια του Μάστριτ και επομένως θα πρέπει να γίνει δεκτή στη ζώνη του ευρώ. Αυτό νομίζω είναι ένα χαρμόσυνο νέο. Επίσης, είναι και ένα θαυμάσιο μήνυμα μήνυμα ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχει διεύρυνση της ζώνης του ευρώ. Επίσης, είναι θετικό μήνυμα αυτό για όλα τα κράτη της Βαλτικής Ζώνης, γιατί αυτό τι σημαίνει, ότι η ζώνη μπορεί να κάνει και μεταρρυθμίσεις και να προωθήσει σωστές πολιτικές. Είναι καλό μήνυμα και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Μήνυμα που λέει ότι όταν σεβόμαστε τα κριτήρια του Μάστρεκτ, το βραβείο είναι η προσχώρηση στην Ευρωζώνη. Τώρα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τακτοποιήσουν τις πολιτικές τους, τον προϋπολογισμό τους και τα δημοσιονομικά τους, ούτως ώστε ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη. Το παράδειγμα της Εστονίας είναι ένα καλό παράδειγμα. Είναι παράδειγμα ότι υπάρχει δυνατότητα για δημοσιονομική πειθαρχία, ακόμη και στις συχνές αγελάδες. Ο κύριος Κούτας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην αρχή της ε, κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι βαλτικές χώρες ε, από τίγρης ε, έγιναν ασθενείς. Τώρα όμως, μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο, η Εστονία ετοιμάζεται να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Θα ενδυναμώσει αυτό την Ευρωζώνη σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι καλό που η Εστονία αποφάσισε να προχωρήσει στην ένταξη αυτή και που ξεπέρασε την κρίση χάρη στα κατάλληλα μέτρα. Τα, οι βαλτικές χώρες έχουν χαμηλό δημόσιο χρέος ε, που αυξάνει την ευελιξία τους σε περίπτωση που χρειαστούν εξωτερικό δανεισμό. Ε, ο λόγος μεταξύ δημοσίου χρέους και ΑΕΠ είναι 7,2% στην Εστονία. Κάτι που είναι πολύ πολύ πιο κάτω από το μέσο κοινοτικό όρο. Θα πρέπει να μάθουμε και να διδαχτούμε από την Εστονία και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ της σύνεσης και της λιτότητας. Παρά τα στοιχεία αυτά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τις κοινωνικές ε, συνιστώσεις ε, από την υιοθέτηση του ευρώ. Υπάρχει κίνδυνος αύξηση των τιμών και ελπίζω ότι οι εστονικές αρχές θα καταφέρουν να εφαρμόσουν ε, ισορροπημένες ε, δημοσιονομικές πολιτικές, ώστε οι θυσίες να μην πάνε χαμένες. Οι συνάδελφοί μας μίλησαν για τον κίνδυνο του πληθωρισμού επίσης. Τελευταίο και σημαντικό, η υιοθέτηση της, ε, του ευρώ από την Εστονία έχει και συμβολική αξία. Συμβολική αξία για τις ανατολικές χώρες που δεν είναι και τόσο πρόθυμες αυτές τις εποχές κρίσης να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Ε, ένα λεπτό, Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, χαρητήρια στην Εστονία. Στην Ευρώπη έχουμε πολλά προβλήματα και νομίζω ότι ακριβώς εκεί χρειαζόμαστε βοήθεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στην Ευρώπη, όπως είναι η Εστονία. Κάποιοι όμως απλά περιμένουν έτσι λίγο διστακτικά, ε, φοβισμένοι, να περάσει αυτή η κρίση, όπως η χώρα σας, η χώρα μου, όπως η Δανία. Νομίζω ότι εδώ οι ιδρυτές πατέρες της Ευρώπης με τον ίδιο τρόπο θα είχαν αντιδράσει. Κάπως έτσι ξεκίνησε η Ευρώπη. Κυρία Πρόεδρε, σε περίοδο κρίσης η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί. Όταν είμαστε περισσότεροι, είμαστε και πιο ισχυροί. Ισχύς εν τη ενώση, όπως λέμε. Πρέπει να υπάρχει μια Ευρώπη ενωμένη και που να προβάλλεται. Μπράβο, μπράβο, μπράβο λοιπόν στην Εστονία. Ευχαριστώ. Τώρα περνάμε λοιπόν στη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Μπασέσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Εσθονία για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να τηρήσει τα κριτήρια σύγκλησης και θέλω να τη συγχαρώ και για τις σόφρονες πολιτικές που ακολουθεί. Γίνεται λοιπόν η Εστονία 17η χώρα που υιοθετεί το ευρώ σε μια δύσκολη περίοδο για την ευρωπαϊκή οικονομία, όταν αυξάνεται η κερδοσκοπία και όταν αυξάνονται και ανησυχίες εξόδου για έξοδο πιθανή κάποιων χωρών από την ευρωζώνη. Άρα το μήνυμα της Εστονίας είναι πολύ ισχυρό για μια ενδεχόμενη διεύρυνση ε, της ζώνης του Ευρώπης Ανατολάς. Έγιναν διάφορες αναλύσεις, έγιναν κάποιες ε, εκτιμήσεις και για τη Ρουμανία για το 2009. Βλέπουμε ότι δεν τηρεί πληρεί όλα τα κριτήρια για ένταξη στην Ευρωζώνη. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν το ευρώ να το υιοθετήσουν μόνο όταν είναι πλήρω έτοιμα γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυβέρνηση και τον εστονικό λαό η Λιθουανία ήταν σε αυτή την ε, πορεία πριν από λίγα χρόνια, αλλά της έλειψαν ε, κάτι δεκαδικά για την εισαγωγή του ευρώ. Είμαστε διαφορετικοί. Πήραμε διαφορετικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές της πορείας μας. Η Ιστονία είχε μια άλλη στάση, πήρε λιγότερο δημογωγικές αποφάσεις και πρόχθησε συνετές πολιτικές σε ό,τι αφορά την οικονομική και φορολογική πολιτική. πιστεύουμε εμείς οι βαλτικές χώρες ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε τα ίδια θετικά αποτελέσματα με την Εστονία. Ακόμα μια φορά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον ε, Υπουργό Οικονομικών που ήταν και παλιός ε, Ευρωβουλευτής που συνεισέφερε τα μάλα για αυτήν την επιτυχία. Συγχαίρω πραγματικά από καρδιά στην κυβέρνηση της Εστονίας που οδήγησε τη χώρα σε αυτή το, την καλή έκβαση. Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο κ. Μπρόνς που μίλησε πριν από λίγα, λίγα λεπτά, ε, είπε αυτά που ήθελε να πει και μετά έφυγε, δείχνει κάποια πράγματα για αυτή την ε, συζήτηση. Ε, το ενδιαφέρον με την Εστονία είναι ότι ε, δίνει ψήφο εμπιστοσύνη. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνη για την Εστονία και ψήφο εμπιστοσύνη για, για το ευρώ. Η πραγματικότητα για την, για την Εστονία είναι ότι χωρίς την πειθαρχία που έδειξε ε, η Εστονία δεν υπάρχει καμία ελπίδα και για τους υπόλοιπους. Ο κύριος Ζάβα. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, δεν θα μπορέσω να συγχωρέσω τον εαυτό μου εάν ε, δεν επωφεληθώ για να συγχαρώ τους Εστονούς συναδέλφους η Εστονία μπόρεσε να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα σε πολλούς τεμούς ε, τομείς τα τελευταία έτη μπόρεσε να αναθεωρήσει τη φορολογία της να αναβιώσει την οικονομία της δεκαετία του 1990 πράγματα και ε, επιτεύγματα τα οποία δεν μπόρεσαν να φτάσουν αλλά άλλες χώρες. Θα είναι ένας ισχυρός εταίρος ή στο ευρώ, θα είναι πολύ προσεκτική και θα συμβάλλουν στη σταθερότητα του, του νομίσματός μας. Και τώρα δίνω το λόγο ε, στον ε, Επίτροπο κύριο Ρέν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για την στήριξη των ε, μελών του Ευρωκοινοβουλίου και θα ήθελα να σας πω για ποιους ε, λόγους υπήρξε τόσο στενό χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση της εκθέσεως Κυκλούνα διότι η ημερομηνία που για την προθεσμία της αξιολογήσεως των στοιχείων για να μπορέσουν να δημοσιευθούν τα στοιχεία αυτά από την Eurostat ήταν ε, περιορισμένη και η, Eurismen, η Eurostat ε, δέχτηκε να ε, επιβεβαιώσει τα φορολογικά στοιχεία ε, πρώτων τακτών ημερομηνιών διότι θέλαμε να εξασφαλίσουμε ένα ποιοτικό προϊόν και δεν θέλαμε να πιέσουμε περαιτέρω την κατάσταση. Αυτό δεν θα το επιτυγχάναμε και δεν θέλαμε να διακινδυνεύσουμε και τα στοιχεία όλων των άλλων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος και ε, της σταθερότητος ε, του Συμφώνου Αναπτύξεως που είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Χρησιμοποίησαμε δηλαδή τα ίδια στοιχεία και τα ίδια θα χρησιμοποιήσουμε και αύριο στην Επιτροπή όταν ε, θα λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τα 16 υφιστάμενα ελλείμματα και τις θέσεις των, των κρατών μελών του ευρώ. Αυτά τα διαδικαστικά στοιχεία λοιπόν οδήγησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία χρειάστηκε να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να συγχαρώ του μέλη της Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων που είχαν αναφερθεί και συζητήσει ήδη τις τις προοπτικές Εστονίας για τη σύγκληση και να ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ανα πάσα στιγμή εξετάζουμε την κατάσταση στην Εστονία. Είναι προφανές ότι η Εστονία πρέπει να παραμείνει και να επαγρυπνά για να μπορέσει να εξασφαλίσει την μακροοικονομική της εξέλιξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί πολύ επισταμένα. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι ελπίζω ότι η Εστονία θα είναι σύμμαχος και θα επιβάλλει την φορολογική πειθαρχία. Χρειαζόμαστε τέτοιους συμμάχους στο ευρώ και γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με την Εστονία για να εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και ε, της, ε, ε, τη βιωσιμότητα της Ευρώπης. Και τέλος νομίζω ότι ο κύριος Μπρόνς αναφέρθηκε ότι υποτιθεμένως η Εστονία θα χάσει την πρόσφατα ανακτηθήσα ανεξαρτησία της. Αλλά ίσως θα έπρεπε να απαντήσω στον κύριο Μπρόντς και να του πω ότι αυτό έχει σχέση με το σκεπτικό το οποίο ακολούθησε ο παππούς μου πριν από 15 χρόνια για ε, το δημοψήφισμα ε, για την προσχώρηση της Φιλανδίας στο ευρώ. Είπε ότι ε, από όταν δεν ήθελα να κοιτώ προς Ανατολάς πάντοτε προσέβλεπα προς δυσμάς. Λοιπόν, Ευχαριστώ και τέλος ο εισηγητής έχει το λόγο. Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Όλη Ρεν για τις εξηγήσεις σας. Καταλαβαίνω το χρονοδιάγραμμα είναι τέτοιο που δεν θα πρέπει να καθυστερήσει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ε, εισηγητές για τις ε, συμβουλές τους και για τις σημαντικές τροπολογίες που υποστηρίζω και ενσωμάτωσα στην έκθεση. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ στον Ήβα Παντάρ που είναι στονός και πρώην υπουργό Οικονομικών καθώς και ο κύριος Γιούγκεν Λίτζι για τις ειλικρινείς εξηγήσει που μου έδωσαν κάθε φορά που χρειάστηκα τη βοήθειά τους. Ε, εύχομαι κάθε επιτυχία στον εσθονικό λαό. Μέχρι στιγμής τα κατάφεραν και διέψευσαν τους επικριτές. Ε, ελπίζω να συνεχίσουν και να επαγρυπνούν για την οικονομία τους, για την ανταγωνιστικότητά της, ούτως ώστε αυτή η επιτυχία θα σημειωθεί και στο μέλλον ε, ως μέλος του, της Ευρωζώνης. Θα ήθελα ε, οι βουλευτές να υπερψηφίσουν αυτή την έκθεση. Αξίζει και είναι σωστή η αίτηση της Εστονίας και όταν ψηφίσει την Τετάρτη το Κοινοβούλιο ελπίζω να επιβραβεύσει την Εστονία και να δείξει ότι μπορούμε να αναζωογονήσουμε την Ευρωζώνη. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της διάταξης στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού με βάση το άρθρο 150. Ο πρώτος στο κατάλογό μου είναι η